Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε την απογευματινή μα σύνοδο με τα προβλεπόμενα σημεία στην ημερήσια διάταξη. Το πρώτο θέμα είναι τα πρακτικά της χθεσινής και της σημερινής πρωινής συνεδρίαση; Αν μέχρι την γνωστή προθεσμία δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, θα θεωρηθούν συγκεκριμένα τα πρακτικά. Παίρναμε στα κατεπήγοντα τώρα συζητήσεις επί περιπτώσεων παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτου δικαίου. Πρώτο θέμα είναι η Μαδαγασκάρη. Και ο πρώτος έχει το λόγο ο κύριος Τσάρλ Στάνοκ. Πρόεδρε, πριν από έξι χρόνια η παράνομη κυβέρνηση του Μεχαβασκάρης που, χαρακτηρίζεται από καταχρήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, βγήκε και υποσχέθηκε ότι θα έπαιρναν τέλος η παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο. Αλλά Πολλοί από τους ε, κατοίκους της Μαγαδασκάρης ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν συγκεκριμένα στοχευμένα μέτρα κατά του Ρανζολίνα. Και είναι βασικό να εφαρμοστούν οι συνθήκες, οι όροι της συνθήκης του Κοτονού και να εφαρμοστούν κυρώσεις. Η Αφρικανική Ένωση θα μπορούσε να κάνει πολλά πιο πολλά. Και είναι λίγες ε, οι συγκεκριμένες δράσεις που έχουν αναλευτεί. Θα πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ Ρατζολίνα και τον, να επιστραπεί στον πρώην πρόεδρο να επιτραπεί στη Μαγαδασκάρη. Ο Ρατζολίνα επίσης θα πρέπει να επιτρέψει στους αντιπάλους του να συμμετέχουν στις προεδρικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Αλλά δυστυχώς ε, η, η, η δεν είναι καλή για τη Μαγατασκάρη. Ελπίζω τους επόμενους μήνες τα πράγματα να επιληθούν και μάλιστα με τρόπο. Σας ευχαριστώ. Επόμενο σομιλητής. Η κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε στην Ολομέλεια το δράμα της Μαδασκάρης. Από το ψήφισμά μας του Φεβρουαρίου του 2010 και μέχρι σήμερα, δυστυχώς ε, τα πράγματα όχι μόνο δεν έχουν βελτιωθεί, αλλά έχουν επιδεινωθεί για το λαό της Μαδασκάρης. Και η σκέψη μου στρέφεται ακριβώς προς αυτό το λαό, γιατί αυτός ο λαός είναι το πρώτο θύμα αυτής της κατάστασης. Πέραν τούτου γίνεται και μία πάλι για την εξουσία αυτή τη στιγμή που φαίνεται ότι είναι ατέρμονη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ε, εδώ και ένα χρόνο ε, διατρανώσει την υποστήριξη του ε, σε μια δημοκρατική διαδικασία που θα οδηγήσει στην διεξαγωγή εκλογών. Κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμη μέχρι σήμερα. Ο Ρατζολίνα εξακολουθεί να βρίσκεται στην εξουσία και δεν δικαιούται να είναι υποψήφιος στις νέες εκλογές. Αυτό το υπενθυμίζουμε και στο τωρινό μας ψήφισμα. Θα ήθελα όμως εδώ να απευθύνω έκκληση ώστε οι διαπραγματεύσει που συνεχίζονται στην κοινότητα με συμβουλή Αφρική ΑΝΤΚ και που δεν έχουν ευοδοθεί μέχρι σήμερα να συνεχιστούν και να έλθουν σε αίσιο πέρα. Σήμερα υιοθετώ ένα πιο μετριοπαθέ ύφο. Ακριβώ γιατί πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μια ευκαιρία στι διαπραγματεύσει που πρέπει να γίνουν κάτι επιγόντω και ευελπιστώ ότι θα ευοδοθούν και όλα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Δεκάιζερ. Ο επόμενος είναι η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σήμερα η Γκουε δεν μπορεί παρά να εκφράσει τη λύπη της για το ύφος των ψηφισμάτων. Το ίδιο Βέβαια αυτό δεν ισχύει για τη, ισχύει και για τη Μαδαγασκάρη. Το 2010 το είχα καταγγείλει στο προηγούμενο καταπήγον ψήφισμά μας. Στη Μαδαγασκάρη αλλά και σε άλλες αφρικανικές χώρες η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει την πολιτική της ανημπορία. Και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην προσπάθειά μας με αναστολή των, της αναπτυξιακής βοήθειας να επηρεάσουμε τα πράγματα, γιατί το μόνο θύμα του μέτρου αυτού θα είναι ο λαός Μαδαγασκάρης. Πραγματικά δεν φταίει σε τίποτα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε το διαμέσο λαβητή της κοινότητας ανάπτυξης Μεσημβρινής Αφρικής που εδώ και ένα χρόνο ε, έχει άοκνες προσπάθειες για να βρει μια λύση. Θα προσπαθούσαμε ε, να συγχαρούμε και τον κύριο Σισάνο που υπέβαλε ένα οδικό χάρτη στην κοινότητα ανάπτυξη Μεσηβινή Αφρική για τη διέξοδο από την πολιτική κρίση στη Μαδαγασκάρη. Το Σάββατο θα γίνει στο Johannesburg μια νέα διάσκεψη κορυφή τη ΑΝΤΕΚ και ελπίζουμε και οι εμπλεκόμενε πλευρέ τη Μαδαγασκάρη να εγκρίνουν τον οδικό χάρτη. Θα θέλαμε να πούμε στο λαό τη Μαδαγασκάρη ότι αυτό θα πρέπει να επιλέξει την κυβέρνησή του χωρί διεθνή πίεση. Στο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να του βοηθήσει δεν θα εγκρίνουμε αυτό το μεροληπτικό ψήφισμα που αντί να υποστηρίξει τις την κοινότητα ανάπτυξης ε, της Μεσημβρινής Αφρικής ρίχνει λάδι στη φωτιά και με, την, ε, με τις κυρώσεις επιδεινώνει την κατάσταση. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως και οι προλαλήσαντες συνάδελφοί μου και εγώ πρέπει να διαπιστώσω ότι ήδη από το Φεβρουάριο του 2010, δηλαδή από τη στιγμή που συζητήσαμε για πρώτη φορά την κατάσταση στη Μαδαγασκάρη, δεν έχουμε καμία ε, θετική εξέλιξη. Μπορούμε να πούμε επομένως ότι δεν έγινε η μετάβαση προς την δημοκρατία. Μάλλον ε, υπάρχει μετάβαση προς μια κατάσταση χειρότερη από αυτήν που ε, διαπιστώναμε την προηγούμενη, την προηγούμενη χρονιά. Η συνεδρίαση της CADC, ε, της Κοινότητας Ανάπτυξης ε, της Μεσημερινής Αφρικής, ε, φαινόταν ότι θα έχει κάποια καλή εξέλιξη και ελπίζομαι ότι και η συνάντηση αυτή, αυτού του Σαββάτου θα έχει κάποια θετικά αποτελέσματα. Όμως είναι γεγονός ότι έχει επιδεινωθεί ιδιαιτέρως η κατάσταση στην Μαδαγασκάρη. Οι άνθρωποι εκεί ζουν με λιγότερο από ένα δολάριο την ημέρα. Χρειαζόμαστε ένα ουδέτερο, συνενετικό και αποφασιστικό καθεστώς μετάβασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά το πραξικόπημα και με την κυβέρνηση του Ρατζολίνα, η Μαδαγασκάρη έχει μετατραπεί σε ένα πόλο πολιτικής αστάθειας χωρίς διάκριση εξουσιών, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ελέγχονται από την κυβέρνηση με κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρήση βίας ε, των αρχών ε, ασφάλειας εις βάρος του, λαού, του άμαχου πληθυσμού που υφίσταται τις συνέπειες αυτής της κατάστασης. Η χώρα δεν έχει σημαντικούς πόρους και τους λείπουν και νερό, βασικά τρόφιμα, υγειονομικές υπηρεσίες, παιδεία, υγεία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει την παροχή ανθρωπιστική βοήθεια προ το λαό τη Μαδαγασκάρη και θα πρέπει να συμβάλλει στην ανέβρεση συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών που να διευκολύνουμε μια ουδέτερη, συνενετική, μεταβατική κυβέρνηση προκειμένου να επανέλθουμε στη συνταγματική τάξη και να ε, διεξαχθούν ελεύθερες, δημοκρατικές και διαφανείς εκλογές με συμμετοχή όλων των πολιτικών κινημάτων και πολιτικών ηγετών με ελεύθερο τρόπο, ώστε να μπορέσει ο λαός της Μαδαγασκάρης να αποφασίσει από μόνος του για το μέλλον του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Για μία ακόμα φορά καταδικάζει η ομάδα των Πρασίνων τον τρόπο με τον οποίο ε, ανέλαβε την εξουσία στην Μαδαγασκάρη ο κύριος Ροζοελίν. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά την κοινωνική κατάσταση, οι παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε πρόκειται για ε, καταχρηστική μεταχείριση των μέσων ενημέρωσης, είτε πρόκειται για καταχρηστική μεταχείριση πολιτών, παράνομες κρατήσεις κλπ. Είναι πολλές. Οι ηγέτες τη ε, της βρίσκονται στη φυλακή και απαιτούμε την ε, απελευθέρωσή τους. Ε, επίσης, οι φυσικοί πόροι ε, της χώρας απειλούνται και επίκειται μεγάλη οικονομική καταστροφή. Υπάρχει λαιλάτιση των δέντρων, κυρίως του ροδόδεντρου η κατάσταση είναι τραγική, χρειάζονται άμεσες διαφανείς και δημοκρατικές εκλογές με την βοήθεια της διεθνούς κοινότητας γενικά και ειδικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα ομιλητές από τις ε, πολιτικές ομάδες, ο κύριος Κατσμαρέκα από το ε, ΕΛΚ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, στο ψήφισμά μας στυλιτεύουμε την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την υπερβολική χρήση βίας των αρχών ασφαλείας στις βάρος του λαού. Θέλουμε να βρεθεί πολιτική λύση με σεβασμό των ανθρωπίνων πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων του λαού της Μαδαγασκάρης και επαναφορά στο κράτος δικαίου. Επίσης, δούμε απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και δυνατότητα επαναπατρισμού των πολιτικών εξορίστων. Θέλουμε επίσης επάνωδο της συνταγματικής τάξης στη Μαδαγασκάρη, κάτι που είναι απαραίτητο για να διοργανωθούν διαφανείς, ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές υπό την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής κοινότητας, με δημοκρατικές προδιαγραφές. Βέβαια το δίλημά μας είναι πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον λαό της Μαδαγασκάρης, ενώ δεν αναγνωρίζουμε την κυβέρνηση, το καθεστώς της Μαδαγασκάρης. Πιστεύω ότι παρόλα αυτά μπορούμε να βοηθήσουμε το λαό της Μαδαγασκάρης και υπό αυτούς τους όρους. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρέτσου, εκ μέρους των Σοσιαλιστών Δημοκρατών. Πρόεδρε, δύο χρόνια έχουν περάσει από τότε που έγινε το πραξικόπημα στη Μαγατασκάρη από ένα στρατιωτικό καθεστώς που δεν έχει εκπληρώσει τις υποσχέσεις του σε ό,τι αφορά τη μετάβαση στη δημοκρατία. Η Αφρικανική Ένωση έχει αναστείλει την ε, συμμετοχή της χώρας στους κόλπους της και έχει οδηγηθεί σε διεθνή απομόνωση η κυβέρνηση και ο λαός της Μαγαδασκάρης ε, δεν απολαμβάνει πλέον της διεθνούς προστασίας και βοήθειας. Αυτά στριτεύουμε στο ψηφισμά μας. Θα πρέπει τα μέτρα τα οποία εγκρίθηκαν από την Αφρικανική Ένωση να αναθερεθούν και να βοηθηθούν οι πολίτες της Μαγαδασκάρης πολιτικώς. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιμείνει προκειμένου τα κόμματα στη Μαγαδασκάρη να υπερβούν τις ε, αντιπαλότητές τους και να συμφωνήσουν με τις χώρες της Αφρικανικής Ένωσης πώς θα ξεπεραστεί η κρίση. Θα πρέπει ο πρώην πρόεδρος να επιτρέψει στη χώρα του και να ληφθεί υπόψη ότι δεν είναι δυνατόν να έχει αυτές τι ευκαιρίες μόνο για την υπόλοιπη ζωή του. Ευχαριστώ. Η κυρία Ογιουλάντ, εξ ονόματο των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα πραξικόπημα στην ε, Μαγαδασκάρη ακολουθήθηκε από διαρκή ε, παραβίαση των ανθρωπίων δικαιωμάτων και είδαμε την συγκέντρωση της ε, εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας μαζί με την, τα μέσα ενημέρωση στα χέρια του Ρατζολίνα. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν έχουν αναγνωρίσει αυτή την ε, παράνομη ε, κυβέρνηση. Δεν θα πρέπει ποτέ να αναγνωρίζεται μια τέτοια κυβέρνηση με επίσημες ε, διαπραγματεύσεις και επίσημες σχέσεις, παρά το γεγονός ότι το έχουμε κάνει αυτό στο παρελθόν. Παρά το γεγονός ότι έχω καλέσει την εθνική κοινότητα να προωθήσει μία σαφή μετάβαση προς τη δημοκρατία. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέη, επόμενη μιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Μετά από το πραξικόπημα ε, του 2009 ακολούθησαν πολλαπλές παραβιάσεις ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και ο εγκλισμός στη φυλακή των πολιτικών υπευθύνων της αντιπολίτευσης. Οι πραξικοπηματίες θα πρέπει να τιμωρηθούν, θα πρέπει να βοηθηθούν ο λαός της Ματαγασκάρης να βοηθηθεί έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρεθεί κάποια λύση και να οδεύσει προς την δημοκρατία οι ε, στρατονομίες ε, θα πρέπει να καταργηθούν ε, και θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να σταματήσουν αυτές οι καταχρηστικές μεταχειρήσεις κατά του, πολιτισμού, του πληθυσμού. Συγγνώμη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει νόμιμη συνταγματική εξουσία η οποία θα είναι αποδεκτή από τον κόσμο. Ζητώ από το Συμβούλιο να εντείνει τις προσπάθειες, να επιταχύνει τις προσπάθειες έτσι ώστε να εξευρεθεί η λύση για την ε, ε, άμεση ε, σύγκληση εκλογών. Ο κύριος Ρέπο. Κύριε Πρόεδρε. Η Μαδαγασκάρη είναι η τέταρτη σε μέγεθος νήσος του κόσμου και ο πληθυσμός της έχει πολύ υποφέρει κυβερνάται αυτή τη στιγμή από μια κυβέρνηση η οποία δεν αποτελεί αποτέλεσμα ελεύθερων εκλογών. Οι ε, φυσικοί της πόροι κατασπαταλούνται και μάλιστα υποχρεούται ο πληθυσμός της Μαδαγασκάρης να ζήσει σε απάνθρωπες ε, ε, συνθήκες και στην απόλυτη φτώχεια καταχρηστικές ε, παραβιάσεις, ε, καταχρηστικοί ε, φυλακισμοί, λαιλασία των φυσικών πόρων, των δασών και άλλων φυσικών πόρων της χώρας είναι καθημερινή κατάσταση. Βασανιστήρια καθώς επίσης και εξαφανισμοί ανθρώπων είναι στην καθημερινή ημερήσια διάταξη Βλέπουμε επίσης ε, ότι ε, η χλωρίδα και η πανίδα υποφέρουν παρότι πρόκειται για εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα και πανίδα σε αυτή την περιοχή του κόσμου. Θα πρέπει να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις προσπάθειες του λαού της Μαδαγασκάρης. Ευχαριστώ πολύ. Και ο κύριος Κέλλη. η κατάσταση στην ε, Μαδαγασκάρη είναι μια κλασική κατάσταση, μια κλασική περίπτωση όπου το καλύτερο δεν είναι, ε, το νεότερο δεν είναι καλύτερο από το παλαιότερο τα πράγματα δεν έχουν ε, αλλάξει και τα, οι παλιές κακές συνήθειες ε, παραμένουν. Βλέπουμε βασανιστήρια πνευματικά, ψυχολογικά και ε, φυσιολογικά. Βλέπουμε μεγάλη αύξηση της καταχρηστικής φυλάκισης των πολιτών και βλέπουμε επίσης τον πληθυσμό που ζει με λιγότερο από ένα δολάριο κάθε ημέρα. Θα πρέπει να οργανωθούν ελεύθερες εκλογές ε, έτσι ώστε να υπάρξει νέα κυβέρνηση σε συνεργασία βεβαίως με άλλους ε, διεθνείς οργανισμούς, κυρίως ε, σε συνεργασία με την Αφρικανική Ένωση. Θα μπορέσουμε ενδεχομένω να βοηθήσουμε την χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Η διαδικασία Catch the Eye τώρα. Η κυρία Νασάη θέλει το puhemies, vuoden 2009... Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μετά τις ε, πολιτικές αλλαγές ε, που έλαβαν χώρα στη Μαδαγασκάρη, διαπιστώνουμε μια πολιτική αστάθεια και μια επιδείνωση της κατάστασης. Γινόμαστε μάρτυρες κατάφορης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή και οι χώρες ΑΚΕ συμφώνησαν ότι η Μαδαγασκάρη είχε ανάγκη από μια προσωρινή κυβέρνηση. Νομίζω ότι πλησιάζουμε στο πέρας αυτής της κρίσης χάρη στη συνεργασία τη ΑΝΤΕΚ, τη κοινότητα ανάπτυξη με τη Ιβρινής Αφρική που κάλεσε τα αντίπαλα μέρη να έρθουν στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Τρεις, τρία κόμματα της αντιπολίτευσης αρνήθηκαν να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσεις, κάτι που δίνει την ευκαιρία στο Ρατζολί να συνεχίσει την παραμονή του στην εξουσία παρά τα προβλήματα που δημιούργησε. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει η διεθνή κοινότητα να παρέμβει, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να αφήσουμε να συνεχίζει να κρατά την εξουσία η παράνομη κυβέρνηση του Ρατζολίνα. Κυρία Έδιγκερ Ντεότεμπεργκ, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αιτία της παρούσης πολιτικής κρίσης στη Μαδαγασκάρη ήταν το στρατιωτικό πραξικόπημα που εξανάγκασε πριν από δύο χρόνια σε παρέτηση και εξαιωρία τον εκλεγμένο με δημοκρατικές διαδικασίες πρόεδρο της Μαδαγασκάρης Μάρκο Ραβαλομανάνα. Η ανάληψη της εξουσίας από το στρατό φυσικά στυλιτεύτηκε από την ε, παγκόσμια κοινότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που ανέστηλε αμέσω την αναπτυξιακή της βοήθεια. Παρόλο και επίση η Μαδαγασκάρη απεπέμφθη από την κοινότητα ανάπτυξη Μεσηβρινής Αφρικής και από την Αφρικανική Ένωση, κάτι όμως που οδήγησε σε μεγαλύτερη απομόνωση του νησιού. Η πολιτική κρίση στη Μαδαγασκάρη φτάνει σε ένα οριακό σημείο, αλλά δημιουργείται ταυτόχρονα και μια ευκαιρία οι συνεχεί διαπραγματεύσει μεταξύ των πολιτικών αρχηγών να έρθουν σε αίσιο πέρα. Είναι μια κατάλληλη ευκαιρία να επανέλθουμε στη συνταγματική τάξη και να διοργανωθούν νέε εκλογέ οι συζητήσεις αυτές έχουν μεγάλη σημασία για την επιστροφή των κονδυλίων στη χώρα αυτή που ε, έχασε μέχρι στιγμής 600 εκατομμύρια ευρώ στα πλαίσια αναπτυξιακής βοήθειας εξαιτίας της Ανατολής της. Ελπίζω ότι οι αντίπαλες πλευρές θα καταφέρουν να εφαρμόσουν τον οδικό χάρτη που θα επιτρέψει μεταβατική κυβέρνηση και διεξαγωγή νέων έντιμων και δίκαιων εκλογών. Ο κύριος Φερέιρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τη λύπη μου για την ε, μεγάλη καθυστέρηση της μετάφρασης όλες τις γλώσσες των ψηφισμάτων. Ε, μερικέ ψηφίσματα και προτάσεις δεν τι έχω καν ακόμα στα πορτογαλικά και θα ήθελα να εκφράσω την έντονη διαμαρτυρία μου για την καθυστέρηση αυτή. Θα πρέπει η διεθνή ε, κοινότητα να βοηθήσει μια διαδικασία μετάβαση και επανασυμφιλίωση στη Μαδαγασκάρη, χωρί όμω. Ε, παρέμβαση και παρεμβολή στα εσωτερικά τη χώρα. Θα πρέπει να αφήσουμε το λαό τη Μαδαγασκάρης να αποφασίσει από μόνο του. Είναι προ το συμφέρον του λαού τη Μαδαγασκάρης και όχι προ το συμφέρον των αντίπαλων μερών να συμμετέχουν στι διαπραγματεύσει όλε οι δυνάμει. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις προσπάθειες της κοινότητας ανάπτυξης Μεσημερινής Αφρική για την επίλυση τη σύγκρουση και την ανέβρεση μια πολιτική λύση για διέξοδο από την κρίση. Εμεί θα θέλαμε να διατρανώσουμε την ανάγκη ε, να σεβαστούμε την ικανότητα του λαού της Μαδαγασκάρης να επιλέξει και να προσδιορίσει το μέλλον του. Οκ, okay, θα δούμε τι έγινε με τις πορτογαλικές μεταφράσεις και γιατί καθυστέρησαν τώρα. Επόμενη ομιλήτρια, κυρία Μπασέσκου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα κρίση στην Μαδαγασκάρη αντιπροσωπεύει μεγάλο κίνδυνο για την ε, δημοκρατία και <clears throat> για την ε, ε, σταθερότητα στην περιοχή. Έχει επιτείνει την ανασφάλεια και την βία η πραξικοπηματική ανατροπή του προηγουμένου Προέδρου. Θα πρέπει να δοθεί μια ανακούφιση στον πληθυσμό αυτού του νησιού. Ένα νησί το οποίο αντιμετωπίζει φτώχεια κατά 80%. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αρθούν οι τελωνιακοί δασμοί για την εισαγωγή κλωστοϊφαντουργικών προϊόντων από την Μαδαγασκάρη. Ε, <clears throat> καλωσορίζω τις προσπάθειες της κοινότητας ανάπτυξης της Μεσημβρινής Αφρικής ε, για την επιστροφή της δημοκρατίας στην Μαδαγασκάρη και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εμπλακεί στην αναζήτηση λύσης στο πρόβλημα της Μαδαγασκάρης. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κούτος για να παραμείνουμε στην ίδια γλώσσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η πολιτική κρίση της Μαδαγασκάρης οδήγησε το νησί αυτό σε απομόνωση από την ε, διεθνή σκηνή. Ε, και μετά από ψήφιμα της, των Ηνωμένων Εθνών ε, σταμάτησαν οι βοήθειες που εδίδονται ε, στην Μαδαγασκάρη και υπό τον πρόεδρο Ρατζοελίνα είναι υπό αμφισβήτηση η μετάβαση στη δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα θα γίνουν ακόμα σημαντικότερα εάν σταματήσει η υποστήριξη Προ την Μαδαγασκάρη και θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε την ε, στήριξή μα προς το νησί αυτό και όχι μονάχα ε, λέγοντας ότι θα πρέπει να γίνουν ελεύθερες εκλογές αλλά και με πιο συγκεκριμένου τρόπους. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σιλβέστρα, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, από τον Ιούνιο του 2003 η Μαδαγασκάρη είχε ξαναρχίσει να συμμετέχει ενεργά ε, σε την πολιτική ζωή της Αφρικής. Μετά όμως οι πολιτικές επιλογές ε, την οδήγησαν στους ε, μη, στους μη στους ανεξάρτητους κομμουνιστές. Βλέπουμε ότι 19 μήνες μετά από το πραξικόπημα 8 εκατομμύρια κατοίκων της Μαδαγασκάρη Μαδαγασκάρης ε, δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν ελεύθερα και επομένως μήπως θα μπορούσατε λίγο να μιλάτε με αργότερο ρυθμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, και μετά από αυτές τις ε, εκλογές δεν έσβησε, συγγνώμη, έσβησε κάθε ελπίδα για ελεύθερες εκλογές και δημοκρατικές διαδικασίες σε αυτήν την παλιά απικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε ότι και σε επίπεδο οικονομικό και σε επίπεδο ανθρωπιστικό και κοινωνικό τεράστια είναι η απόσταση που ξεχωρίζει, που χωρίζει μάλλον τους ε, πολίτες της Μαδαγασκάρης ε, από τους υπόλοιπους κατοίκους της Αφρικής. Ε, έχουν ληφθεί αποφάσεις αρνητικές προς την Μαδαγασκάρη και από την Παγκόσμια Τράπεζα και τα Ηνωμένα Έθνη. Θεωρούμε ότι άμεσα με επίγοντα τρόπο θα πρέπει να διοργανωθούν ελεύθερες δημοκρατικές εκλογές στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Διαδικαστικό. I Νταφ για διαδικαστικό και τρέφω απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό σας κύριε Πρόεδρε. Φυσικά ο κάθε ομιλητής επιλέγει την ταχύτητα με την οποία θα εκφωνήσει την ομιλία του. Αναπόκειται στη διακριτική του ευχέρεια. Οι ομιλητές, οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να υφίστανται τις ε, συνεχείς διακοπές του Προέδρου επειδή οι διερμηνεί δεν μπορούν να του προλαβαίνουν. Αυτό θα ήθελα να το πω. The large extents, I agree with you. Σε κάποιο βαθμό συμφωνώ μαζί σας, αλλά δεν μπορώ να γνωρίσω ε, την ε, διαμαρτυρία των διερμηνέων σε περίπτωση που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το ρυθμό. Φυσικά όταν ε, διακόπτω έναν ομιλητή, του επιμετρώ αυτό το χρόνο της διακοπής, ώστε όλοι να είναι ικανοποιημένοι και ο ομιλητής που δεν περικόπηκε και ο χρόνος του και εσείς που ακούτε την ομιλία πολύ πιο ολοκληρωμένη εφόσον γίνεται σε κανονικό ρυθμό, αλλά και των διερμηνέων που μπορούν και την προλαβαίνουν. Νομίζω ότι έτσι μένουμε όλοι ικανοποιημένοι. Ωραία και δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Κορχόλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε από το πραξικόπημα του Μαρτίου η πολιτική αστάθεια στη χώρα αποτελεί κάτι το καθημερινό για τους πολίτες της Μαγατασκάρης. Λόγω της πολιτικής κρίσης έχουν όλο και πιο μεγάλα προβλήματα να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, σε υπηρεσίες οικονομικής περίθαλψης. Αυτοί που έχουν την εξουσία ε, εξουσιάζουν επίσης και την αστυνομία, κατέχουν και τα μέσα ενημέρωσης ε, στρέφονται με βία κατά των πολιτών και οι πρώην πολιτικοί ηγέτες της χώρας έχουν εξαναγκαστεί σε εξορία. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε τη συνταγματική ελευθερία στην χώρα αυτή. Αυτό σημαίνει ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει βοήθεια προς τη Δασκόρη προκειμένου να εξευρεθεί πολιτική λύση. Θα ζητήσω τώρα από τον Επίτροπο, λέει ο Πρόεδρος, να σχολιάσει. Κύριε Οτινιέρ, ποια είναι η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εκπρόσωπος Άστον ε, είναι ιδιαίτερα ανήσυχη για την κατάσταση στη Μαγατασκάρη. Λέμε λοιπόν, βλέπουμε το λαό της όμορφης αυτής ε, χώρας και του ευχόμαστε ε, κουράγιο. Βλέπουμε ποια είναι η πολιτική κατάσταση, ποιες είναι οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά τον πληθυσμό της Μαγατασκάρης που καθημερινά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Εσείς οι βουλευτές ε, και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και προσπαθούμε με διπλωματικές οδούς να ε, δώσουμε ένα τέρμα σε αυτή την κρίση. Εδώ και δύο χρόνια αντιμετωπίζουμε ε, μια δύσκολη κατάσταση και σήμερα βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής στις 7 Ιουνίου πριν από δύο ημέρες λοιπόν έγιναν συνομιλίες μέσα τη κοινότητα ανάπτυξη τη Μεφρινή Αφρική και διαφόρων παραγόντων τη χώρα, προκειμένου να εξευρεθεί μια διέξοδο από την κρίση. Μια οδό ε, η οποία θα βασίζεται στην ε, ουδετερότητα και την αμεροληψία που θα ικανοποιήσει τα συμφέροντα όλων των πλευρών και που θα γίνει αποτεκτή από τη διεθνή κοινότητα αλλά και από τους πολίτες της Μαγατασκάρεξ. Ελπίζουμε οι συνομιλίες να στεφτούν με επιτυχία προκειμένου η Αφρικανική Ένωση και η όλη, το σύνολο της διεθνής κοινότητας συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν την επιστροφή της Μαγαδασκάρης σε μη συνταγματική σταθερότητα την κάθε προσπάθεια μονομερούς ε, κυβέρνησης ε, de facto την απορρίπτουμε. Και γι' αυτό οι Ευρωπαίοι στο Συμβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα συμφώνησαν ε, παράταση κατά έξι μήνες των μέτρων που προβλέπονται στο άρθρο 96 της συνθήκης της του Και από αυτό εξαρτώνται και η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και μέτρων καταπολέμησης της στόχιας. Είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε βοήθεια σε αυτή τη διαδικασία εκδημοκρατισμού και θα πρέπει να βασίζονται αυτά τα μέσα ε, σε έναν οδικό χάρτη ο οποίος θα αποφασιστεί επί τόπου και από τους τοπικούς φορείς και από την κοινότητα ανάπτυξης Μεσημβρινής Αφρικής. περιμένουμε λοιπόν θετικέ εξελίξει μετά από δύο άσχημα χρόνια. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Επίτροπε. Ολοκληρώσαμε τη συζήτηση για τη Μαδαγασκάρη. Η ψηφοφορία θα γίνει περίπου σε μισή ώρα. Δεύτερο σημείο. Το επόμενο σημείο λοιπόν στην ημερήσια διάταξη είναι η επικείμενη απαγγελία θανατικής ποινής στο Γουαντάναμο. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον κύριο